Okay, Καθίστε παρακαλώ, αγαπητοί συνάδελφοι, για να ξεκινήσουμε αυτή την ειδική συνεδρίαση, ανταλλαγή απόψε με τους νέους από την εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή Νεολαία για το ρόλο της εξωτερικής δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των μεταστευτικών ροών. Είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη, ένα τεράστιο ζήτημα και Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολιτικές δυσκολίε και προκλήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει κάποια πολύ καλά πράγματα. Έχουμε χώρε που καλωσορίζουν τους μετανάστες και εργάζονται σκληρά για να εντάξουν ανθρώπου που ουσιαστικά εγκαταλείπουν κάποιες εμπόλεμες ζώνες. Επίση, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δυσκολίε. Χαίρομαι λοιπόν πολύ που θα, θα καλωσορίσω του σημερινού προσκεκλημένου μα. Ε, δεύτερη ε, συναντήσεις τη εκδήλωση Ευρωπαϊκής Νολέας έλαβε χώρα στις 20-21 Μαΐου. Είχαμε 7.000 νέους ανθρώπους που συζήτησαν τις ιδέες τους που παρουσιάζονται σε 10 διαφορετικές επιτροπές στο Κοινοβούλιο. Όλοι οι βουλευτές έχουν λάβει αντίγραφο της έκθεσης της εκδήλωσης για την Ευρωπαϊκή Νεολαία του Μαΐου, του Σεπτέμβριο. Το έγγραφο φέρει τον τίτλο Διαμορφώνοντα στην Ευρώπη 50 ιδέες για το μέλλον». Σήμερα έχουμε τρεις ομιλητές από την εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή Ελέα που θα μας παρουσιάσουν κάποιες ιδέες και κατόπιν θα σα ζητήσω να απαντήσετε στις ιδέες. Θα, ακούσουμε, θα έχουμε λοιπόν τρεις σύντομες παρεμβάσεις από τους βουλευτές ιδίως θα είναι σύντομες οι παρεμβάσεις. Θα δώσουμε το λόγο στους προσκεκλημένους μας, θα ακούσουμε τις ιδέες και θέλουμε τις δικές σας αντιδράσεις σε αυτές τις τρεις ιδέες. Δύο λεπτά για κάθε παρέμβαση το πολύ. Και ελπίζουμε ότι οι ιδέες που θα ακούσουμε από τους ε, καλεσμένους μας σήμερα θα τροφοδοτήσουν την επόμενη συνάντηση για την κοινή έκθεση μεταξύ ε, Επιτροπής ΑΦΕΤ και ΝΤΕΒΕ για τη μετανάστευση. Έχουμε τρεις ομιλητές. Λίντα Σλαπακόβα, οποία είναι αρμόδια διεθνών σχέσεων, ε, είναι εμπειρογνώμονα σε ευρωπαϊκές σπουδές ασφάλειας και ειρήνης και ασχολείται πιο συγκεκριμένα με το θέμα του εξτρεμισμού στην πολιτική ευρωπαϊκής γειτονίας. Έχει εργαστεί στην τσεχική πρεσβεία στις Βρυξέλλες και σήμερα εργάζεται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για τις Πολιτικές Σπουδές. Εδώ έχουμε τη Λίντα και επίσης έχουμε την Αντρέα Γκαβρίλα η οποία ε, έχει λάβει το βραβείο, έχει λάβει μια υποτροφία ε, για το Πανεπιστήμιο του Ντόμ έχει εργαστεί για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, και την ε, Αμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Κογκρέσο και έχει ουσιαστικά εργαστεί ως εθελόντρια ε, για να έχουν πρόσβαση τα θύματα εμπορίας στη δικαιοσύνη. Και Ματέι Τζούσκα, ο οποίος από την Πολωνία μετανάστευσε με την οικογένειά του στη Γερμανία όταν ήταν παιδί, από το 2009 έως το 2015 εργάστηκε στο Γερμανικό Μεταναστευτικό Γραφείο και έγινε πρόεδρος ε, της οργάνωσης νεολαίας της ε, ΣΕΖΗ, της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων και έχει εργαστεί στην ανάπτυξη πολιτικών για τη μετανάστευση. Χωρίς χρονοτριβή, θα δώσουμε το λόγο στη Ματέο με την ιδέα 1 και κατόπιν την Αντρέα για την ιδέα 2 και θα δώσω κατόπιν το λόγο στους συναδέλφους. Παρακαλώ, Ματέους. Ευχαριστώ πολύ. Η πρότασή μου θα επέτρεπε σε όλες τις διπλωματικές αντιπροσωπείες των κρατών μελών της Ένωσης να λαμβάνουν αιτήσει για άσυλο ούτω ώστε να παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια σε όσους χρειάζονται. Θα μπορούν έτσι οι ετούντες να παίρνουν το καθεστώς του ετούντα άσυλο επίσημα ε, χωρίς να ε, δημιουργούνται μποτιλιαρίσματα ε, από το, του, που έρχονται. Μία πρεσβεία μόνο λειτουργεί έτσι. Αυτό θα ήταν μεγάλη αλλαγή, γιατί θα μπορούσαμε να παρέχουμε προστασία στους ζητούντες άσυλο από την αρχή και από την άλλη οι απο, ε, θα κοινοποιούνταν στους ενδιαφερομένους ε, για να γνωρίζουν τι τύχη είχε η αίτηση. Ε, έτσι θα ε, αποθαρρύνονταν πάρα πολύ από το επικίνδυνο ταξίδι μέχρι την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, στο Γερμανικό Γραφείο Μετανάστευσης είδα πολλές φορές ε, ανθρώπους ε, που έλαβαν τη διαβεβαίωση ότι έγινε δεκτή η αίτηση, αλλιώς δεν θα έκαναν το επικίνδυνο ταξίδι. Δεν θέλουμε μια κατάσταση όπου να ε, ε, ε, διακινδυνεύουν και να πεθαίνουν άνθρωποι στο ταξίδι. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι μπορεί οι άνθρωποι να μπορούν να φύγουν από τη χώρα τους για να ε, τηθούν άσυλο. Οι διπλωματικές ε, θα μπορούσαν να, δώσουν ανθρωπιστική βοήθεια και να προωθήσουν τις αιτήσει ασύλου. Έτσι θα μειωθεί η παράνομη μετανάστευση και ο ρόλος των διακινητών. Δεν είναι νέα μορφή ασύλου αυτό, αλλά έχει μακρά παράδοση στη Λατινική Αμερική και τον Καναδά. Ωραία. Και στο χρόνο πολύ ωραία, δύο λεπτά. Ελπίζω οι συνάδελφοι να τηρήσουν επίσης το χρόνο τους. Η Ανδρέα Γκαβρίλα είναι η επόμενη ομιλήτρια που θα παρουσιάσει την επόμενη ιδέα. Η Ανδρέα. Η πρότασή μου σήμερα αφορά τη δημιουργία ασφαλών ζωνών η Ευρωπαϊκή Ένωση στις χώρες ε, όπου υπάρχουν συγκρούσεις αντί για τους καταβλισμούς προσφύγων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, οι καταβλισμοί θα πρέπει να γίνουν πόλεις ασφαλείς με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι ασφαλείς πόλεις μπορούν να έρθουν σε εταιρική σχέση με ευρωπαϊκές πόλεις, αλλά καταρχήν είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν αυτές οι ασφαλείς ζώνες στις χώρες σύγκρουσης με το να υπάρχει στρατιωτική ασφάλεια η οποία πρέπει να γίνει σε συνεργασία με όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και συγχρόνως προσπάθειες της ε, παγκόσμια κοινότητας. Υπάρχει μια δήλωση της διάσκεψης κορυφής της Νέας Υόρκης για τους μετανάστες και πρόσφυγες που υπογράφηκε από πάνω από 190 χώρες για την ανάγκη να επανέλθει η σταθερότητα και η ασφάλεια για τους πρόσφυγες. Επίσης πρέπει να υπάρχουν ευρωπαϊκές συγκεκριμένες δράσεις, να υπάρξουν χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υπάρξει καλύτερη υποδομή υγείας και εκπαίδευσης για τους πρόσφυγες και να δώσει στους ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε αυτές τις πόλεις τη δυνατότητα να αυτοδιακυβερνούνται και να είναι αυτάρκης. Αντί να έχουν σπίτια, να έχουν τα υλικά να φτιάξουν το σπίτι τους. Αυτοί οι οποίοι μένουν προσωρινά σε μια ασφαλή πόλη, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην υγεία και στην παιδεία, αλλά θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν και την προσωπικότητά τους και τη ζωή τους και να γίνουν οικονομικά ανεξάρτητοι βάσει του κράτους δικαίου και χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση ή μπορούν να έχουν ένα μικρό χωράφι να καλλιεργούν. Ευχαριστώ. Έχουμε δύο ιδέες και στην ανάπτυξη, στην Επιτροπή Ανάπτυξης θα μιλήσουμε για τη Συρία σήμερα, για το πώς θα φτάσει στους δικαιούχους η ανθρωπιστική βοήθεια και φυσικά ουσιαστικά θα δούμε και πώς υλοποιείται και η δική σας ιδέα για την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών ε, στο πιτέρισμα της μετανάστασης βοηθά. Τι θα κάνουμε, έχουμε τρία σύνολα ιδεών, έτσι λοιπόν ε, θα το επαναλάβουμε αυτό δύο φορές. Τώρα έχουμε δύο βουλευτές ε, για ε, αυτή τη συγκεκριμένη συζήτηση. Η κυρία Ντεσσαρνές, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Συμφωνώ απόλυτα με την πρώτη ιδέα που δόθηκε. Βεβαίω και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να ανοίξει γραφεία έτσι ασύλου στι χώρε όπου έχουμε πρόσφυγε και ιδίω για του Σύρου πρόσφυγε, στην Τουρκία, στην Ιορδανία, πιο συγκεκριμένα και στο Λίβανο. Είναι αλήθεια ότι δεν ε, είναι λογικό ότι κάποιος μπορεί να ζητήσει το δικαίωμα μόνο αν πληρώσει τους δουλεμπρούς και θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του και τι οικογένειάς του για να έρθει παράνομα στην Ευρώπη, ενώ θα μπορούσαμε να το κάνουμε επί τόπου. 100% συμφωνώ λοιπόν με την πρόταση αυτή και υπενθυμίζω ότι ε, ήρθαν, έφτασαν συγγνώμη, στον Καναδά χιλιάδες άνθρωποι και ουσιαστικά η αίτηση ασυλίου τους εξετάστηκε στις ε, γειτονικέ χώρες της Συρίας. Μπράβο λοιπόν για την πρόταση αυτή. Ευχαριστώ. Αυτό είναι κάτι που είδα όταν ήμουν στην Νότιο Τουρκία. Θα ήταν καλύτερα απευθεία ε, ουσιαστικά να συνεργαστούμε με τους ανθρώπους πριν να ξεκινήσουν μαζικά τα μετανάστευση. Ο κ. Παντσέρη. Ευχαριστώ. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλή αναζήτηση νέων ιδεών και ουσιαστικά φέρνει και μια ευαισθητοποίηση μεταξύ των νέων. Εγώ θα ήθελα μόνο να τονίσω τις δυσκολίες απέναντι ιδέε αυτέ αυτές, να έχουν ιδέες αυτές. Παραδείγματο χάρη ιδέα να χρησιμοποιήσουμε τι διπλωματικέ έδρε. Ε, χρειάζεται να πληρούνται κάποιε προποθέσει που σήμερα δεν φαίνονται να υπάρχουν. Καταρχήν θα πρέπει να ενισχύσουμε τι διπλωματικέ έδρε που σήμερα δεν μπορούν να ανταποκριθούν ε, στο να επιτελέσουν αυτό το καθήκον. Και δεύτερον θα πρέπει να έχουμε μια διαθεσιμότητα των ευρωπαϊκών χωρών να δεχτούν του μετανάστε. Γιατί ακούστηκε το παράδειγμα του Καναδά, είναι όμω μια χώρα, ενώ στην Ευρώπη είμαστε σε πολύ πολύπλοκη κατάσταση και όπως είδατε δεν υπάρχει αλληλεγγύη στην ανακατανομή. Και το τρίτο συστατικό είναι το εξή. Όπως ξέρετε υπάρχουν διάφορα είδη μετανάστευση. Ε, τώρα έχουμε, αν έχουμε μια μεταναστευτική, μια ε, οικονομική μετανάστευση θα μπορούσαμε ε, να το αξιολογήσουμε αυτό, αλλά ουσιαστικά αυτό έρχεται σε αντίθεση με κάποιες χώρες που δεν θέλουν καθόλου τους οικονομικούς μετανάστες. Κάποιοι πιστεύουν ότι πρέπει να τους αφήσουμε σπίτι τους τους ανθρώπους αυτούς, αλλά υπάρχει και ένα άλλο είδος μετανάστευσης, οι άνθρωποι που φεύγουν από διώξεις και από εμπόλεμες περιοχές. Και εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα ε, ουσιαστικά χρονικής οργάνωσης. Δηλαδή ε, δεν είναι ότι μπορούμε να ανοίξουμε ε, ουσιαστικά τη δυνατότητα στη διπλωματικά γραφεία να πάει κάποιος ε, και γιατί οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να φύγουν αμέσως. Τώρα ουσιαστικά θα μπορούσαν να διευκολυνθούν οι άνθρωποι αυτοί, αλλά πρέπει να ενισχυθεί αυτή η ιδέα. Και εγώ νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε αυτά τα συστατικά που σας ανέφερα. Ευχαριστούμε. Είναι, υπάρχουν πολλά πρακτικά θέματα για την εφαρμογή αυτών των πολιτικών. Ας ε, κλείσουμε λοιπόν αυτό το θέμα. Η Ανδρέα θα απαντήσει στους δύο βουλευτές. Νομίζω ότι αφορούν περισσότερο την ιδέα του Ματέους. Εγώ θα απαντήσω για την οικονομική μετανάστευση που είναι μια μακρά αντίδραση, μακροπρόθεσμη δηλαδή και πρέπει να εστιάζει στην πρόληψη. Ευχαριστώ. Ο Ματέους. Ευχαριστώ πολύ και την κυρία Σάρνες που υποστήριξε την ιδέα του ΆΙ και για τον κύριο Παντσέρη, σίγουρα είναι δύσκολο να αναλάβουν οι διπλωματικές αποστολές σε αυτό το καθήκον. Όπως είπα όμως στην ιδέα μου, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να επιμεριστεί αυτό το καθήκον μεταξύ όλων των κρατών μελών. Ε, μία πρεσβεία στη χώρα θα μαζεύει τις αιτήσει για άσυλο και θα τις επιμερίζει. Γι' αυτό χρειάζεται περισσότερο προσωπικό βέβαια, είναι σίγουρο αυτό στην πρεσβεία και χρειάζονται και εκπαίδευση. Αλλά από την άλλη πλευρά αυτό που αναφέρεται ότι ένας άνθρωπος στη Συρία που έχει άμεση ανάγκη όταν ε, υποβάλλει αίτηση ασύλου στις πρεσβείες θα πρέπει άμεσα να παίρνουν κάποιον, εφοδιάζονται με ένα έγγραφο για να μπορούν να εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην ε, βάζουν τη ζωή τους σε κίνδυνο μέσα από επικίνδυνα μονοπάτια. Ωραία, είναι πολύ πρακτική αυτή η ιδέα που ίσως ε, πολιτικά είναι δύσκολο να εφαρμοστεί γιατί είναι δύσκολο να, ε, υπάρχει τόση συνεργασία από τα κράτη-μέλη. Ε, υπάρχουν πολλά προβλήματα, προγράμματα όπου έπρεπε να δεχθούμε μετανάστες ε, από καταβλισμούς που ήταν και εκεί κοντά. Ε, υπάρχει δηλαδή εμπειρία σχετικά με το πώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά. Η, επόμενος, ε, η επόμενη, η Λίντα Σλαπακόβα. Ευχαριστώ κυρία <clears throat> Πρόεδρε. Υπάρχουν χιλιάδες οικογένειες που προσπαθούν να διασχίσουν την Μεσόγειο και αυτή πρέπει να είναι και η κύρια εστίασή μας για να εμποδίσουμε τις μαζικές ροές μεταναστών. Γι' αυτό χρειάζεται ένα πλαίσιο δράση Ευρωπαϊκή Ένωση Μεσογείου για να αντιμετωπίσει τι ανάγκε των ε, ανθρώπων αυτών, των νέων ανθρώπων στι χώρε αυτέ, κυρίω με περισσότερη πρόσβαση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την υγεία, κυρίω το να δώσουμε ευκαιρίε σε αυτού, γιατί η έλλειψη ευκαιριών από του κύριου λόγου τη μετανάστευση, αν δεν αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό, με μακροχρόνια προοπτική θα αναγκαστούν και πάλι να φύγουν αυτοί από τις χώρες, σας, από τις χώρες τους για να βρουν κάποιες ευκαιρίες. Δεύτερον, μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ οργανώσεων των νέων και κοινωνίας των πολιτών στην Ευρώπη και αλλού για να αντιμετωπίσουμε τον βίο εξτρεμισμό και να δώσουμε λύσεις στα προβλήματά τους. Εγώ μπορώ να πω ότι ο βίος εξτρεμισμός και η ριζοσπαστικοποίηση, η άκρα ριζοσπαστικοποίηση οδηγεί σε ε, ακραίες καταστάσεις και ανασφάλεια. Γι' αυτό όλη η διεθνή κοινότητα πρέπει να αντιμετωπίσει τον εξτρεμισμό και τη ριζοσπαστικοποίηση και να σταματήσει τη βία με προγράμματα όπως αυτά που υποστηρίζουν την κοινωνία των πολιτών και αυτό μπορεί να εξαχθεί και στην νότια οχθή της Μεσογείου. Επίσης να δημιουργήσουμε από στελεσματικά προγράμματα επανενσωμάτωσης για τους μετανάστες που γυρίζουν στις χώρες τους, ώστε να γίνουν πιο περιεκτικές τοπικές κοινωνίες και να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο στο οποίο οι νέοι μπορούν να αναπτύξουν δυνατότητές τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Αντρέα Καβρίλα θα μας, φέρει, θα μας δώσει τη δεύτερη ιδέα στο θέμα αυτό. Βασιζόμενοι στην αρχή ότι αν δώσετε, μάθετε κάποιον να ψαρεύει θα ψαρεύει όλη τη ζωή και δεν χρειάζεται να του δίνετε ψάρια, εγώ θεωρώ οι επιτροπές ΔΕΒΕ και ΑΦΕΤ θα πρέπει να φτιάξουν ένα σώμα νέων. Ένα σώμα για την ειρήνη από τους νέους. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να βοηθήσουμε τους νέους να αναπτύξουν στις τοπικές τους κοινότητες τις δικές τους ικανότητες και να ακολουθήσουν την ευρωπαϊκή ατζέντα για την μετανάστευση αυτοί οι οποίοι θέλουν να συμβάλλουν μπορούν να πάνε στις αναπτυσσόμενες χώρες και να δώσουν στον τοπικό πληθυσμό τις δεξιότητές τους για τη γεωργία, για την πράσινη ενέργεια κτλ. Γνωρίζετε ότι μπορεί να φτιάξει κανείς ένα ανεμόμυλο από ένα κατεστραμμένο ποδήλατο, αλλά εγώ το είδα από τα μέσα ενημέρωσης όταν κάποιος στο Μαλάουε έχει φτιάξει ηλεκτρικούς ε, ανεμόμυλους, μάλλον ανεμόμυλους που παράγουν ηλεκτρισμό από απλά υλικά. Είναι απαραίτητο λοιπόν να γίνει αυτό σε τοπικές κοινότητες για να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι συγκρούσεων και να υπάρχουν κέντρα για τους νέους. Θα πρέπει να δοθεί σε αυτούς τους νέους ένα βασικό εισόδημα και χρήματα για την εκπαίδευση σε τοπικό επίπεδο και αυτή η υπηρεσία θα πρέπει να υποστηριχθεί. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να είναι αντικείμενα αναφορών και να γίνουν ορατά για να είναι και ένα παράδειγμα για τους άλλους. Και κυρίως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βοηθήσει τους νέους να έχουν μια ζωή η οποία θα έχει κάποιο νόημα και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθεί ο ριζοσπαστισμός και ο εξτρεμισμός μπορεί να του οδηγήσει στο θάνατο και μόνο. Ευχαριστώ συνάδελφε έχετε κάποιες ε, απαντήσεις σε αυτές τις ιδέες. Εδώ ακούσαμε το, την υποστήριξη των νέων να συνεργαστούν μαζί τους για να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα. Ξέρουμε ότι στην Αφρική η δημογραφική η ανάπτυξη είναι τεράστια πρόκληση σε ό,τι αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασία. Και χθε ακούσαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση στην Επιτροπή Ανάπτυξη για τα μικρά χωριά, πώ τα αφρικανικά χωριά αναπτύσσουν οι άνθρωποι λύσει εκτό δικτύου για την παραγωγή ενέργεια. Και ξέρουμε ότι δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα και πέφτει το σκοτάδι στι 6 το βράδυ. Έτσι λοιπόν και το θέμα τη μεταφορά τεχνολογική γνώση είναι στην υπηρεσία διάταξη. Υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να αντιδράσουν σε αυτές τις δύο ιδέες, κάποιοι βουλευτές. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τις ε, ιδέες σας ε, και που ήρθατε εδώ να μας τις παρουσιάσετε. Να προσθέσω κάτι. Έφτασα καθυστερημένη για τη μουσέλη συνεδρίαση. Ε, ίσως να καλύψατε ήδη αυτό το θέμα όμως. Εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο αγωνιζόμαστε και για πολλά χρόνια, τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια, ζητάμε μία λύση ε, έτσι ώστε να υπάρχουν κοινέ προσπάθειε μεταξύ των κρατών μελών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πριν δύο εβδομάδε ήμουν στη Νέα Υόρκη, είχαμε την πρώτη σύνοδο σε επίπεδο ΙΕ για τη μεγάλη μετακίνηση προσφύγων και μεταναστών. Και φυσικά εκεί συζητήσαμε για μια παγκόσμια προσπάθεια που χρειάζεται να γίνει, γιατί η μετανάστευση και η υποδοχή των προσφύγων είναι παγκοσμία πρόκληση και χρειάζονται φυσικά παγκοσμίες λύσεις, αλλά πόσο αξιόπιστοι μπορούμε να είμαστε ως Ευρωπαϊκή Ένωση όταν ε, εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούμε να έχουμε κοινέ λύσει που χρειαζόμαστε απελπισμένα, γιατί σήμερα έχουμε 6 από τα 28 κράτη-μέλη που μόνα του προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το 80% των αιτήσεων ασύλων που κατατίθεται στην Ευρώπη. Αυτό δεν είναι βιώσιμο για κανέναν. Αλλά όπω σε κάθε προσπάθεια, αν ε, μπορεί να, να την επιμερίσουμε στους 28 θα είναι βιώσιμη για όλους. Αυτό υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι πολύ σημαντικό. Εμείς ως βουλευτές επιστρέφουμε στις πατρίδες μας σχεδόν κάθε εβδομάδα και προσπαθούμε να εξηγήσουμε και προσπαθούμε να ξεκινήσουμε μία συζήτηση με τους συμπολίτε μας στις πατρίδες μας. Δεν είναι πάντοτε εύκολο να κατανοήσει κανείς τις διάφορες ευθύνες μεταξύ Συμβουλίου, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις διάφορες αρμαδιότητες. Όμως πρέπει να επιμείνουμε σε αυτή την επιμερισμένη προσπάθεια γι' αυτό διαφορετικά δεν μπορούμε να το κάνουμε. Οι αναγόμες. Και εγώ λυπάμαι που δεν μπόρεσα να ακούσω όσο υπόθηκαν γιατί ήρθα από μια άλλη συνεδρίαση. Αλλά άκουσα το τέλος των παρεμβάσεων και πραγματικά ε, ήταν πολύ στοχευμένα όσα υπόθηκαν. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τους νέους να είναι ενεργοί και να προωθούν τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό με οδηγεί στον από πω το εξής την ανάγκη ε, πάνδρωσης. Θα πρέπει οι κυβερνήσεις μας ε, να επενδύσουν στρατηγικά σε προγράμματα προκειμένου να καταπολεμήσουν τη διάδοση των εξτρεμιστικών ιδεολογιών που οδηγούν στη βία. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει αρκετή δουλειά από τις κυβερνήσεις μας στον τομέα αυτό. Εμείς σε αυτό το κοινοβούλιο εδώ και πολύ καιρό, πριν ένα έτος, αναφέραμε το θέμα της πρόληψης. Εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ λίγες οι επενδύσεις και οι επενδύσεις αυτές δεν θα λειτουργήσουν αν δεν εμπλακούν και οι νέοι, οι ενώσεις των νέων σε τοπικό επίπεδο προκειμένου να μπορούν να είναι πραγματικοί πρωταγωνιστές για να καταπολεμήσουν αυτή την ιδεολογία των τρομοκρατικών ομάδων που δυστυχώς οδηγεί σε περισσότερη βία. Φυσικά πρέπει να έχουμε και πολιτικές πραγματικά να δίνουν αρμοδιότητες στους νέους και θα πρέπει να υπάρχουν και κοινωνικές ευκαιρίες, δουλειές, γιατί δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να σκεφτόμαστε ότι θα κάνουμε καλή δουλειά και θα έχουμε καλά αποτελέσματα στον τομέα της πρόληψης αν ταυτόχρονα δεν προσφέρουμε βασικές ευκαιρίες στους νέους δηλαδή δημιουργία θέσεων εργασία κτλ. Και ουσιαστικά πρέπει να ξεφορτωθούμε αυτές τις ηλίθιε πολιτικές λιτότητας που υποσκάπτουν και τη δική μας ε, ασφάλεια και θα πρέπει να έχουμε κοινωνική ολοκλήρωση. Επίσης, συμφωνώ με όσο είπε η Έλλη για το θέμα των προσφύγων. Όπως οι κυβερνήσεις μας διαχειρίζονται την εισρωή προσφύγων και μεταναστών δεν θα σταματήσει φυσικά αυτό με φράκτες πολέμους. Θα έρχονται και όλο και περισσότεροι θα έρχονται και ουσιαστικά η Ευρώπη θα πρέπει να όσο μάλλον δεν παρεμβαίνει για την επίλυση της ε, σύραξης τόσο περισσότεροι θα έρχονται. Έχουμε ε, θα πρέπει να έχουμε μία προσέγγιση που δεν θα συνεχίσει να δίνει δουλειά στους δουλεμπορούς. Ε, και ο Αντώνιο Γκουτιέρες είπε ξέρουν ε, οι δουλεύουν πώ να διαχειριστούν την ροή των προσφύγων. Εμεί είμαστε αυτοί που δεν το κάνουμε αυτό, γιατί κατά κάποιο τρόπο ουσιαστικά δίνουμε και βοηθάμε τους ανθρώπους αυτούς ε, να έχουν δουλειά. Ο μόνος τρόπος να σταματήσουμε ε, ουσιαστικά τη δουλειά των δουλεμπόρων είναι να ανοίξουμε νόμιμες και ασφαλείς οδούς για τους ανθρώπους να μπορούν να έρθουν οι άνθρωποι είτε ως πρόσφυγες και να ζητήσουν προστασία είτε ως μετανάστες. Όσο αρνούνται κυβερνήσει κυβερνήσεις να το κάνουμε αυτό, τότε θα δίνουμε δουλειά στους διακινητές και πρέπει οι νέοι να υψώσουν τη φωνή τους και να μιλήσουν γι' αυτό. Ε, δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμη. Να ακούσουμε τις επόμενες δύο ιδέες και μετά να σχολιάσετε στο τέλος, αλλιώς δεν θα προλάβουμε. Πάμε λοιπόν στις επόμενες δύο ιδέες. Δεν ξέρω αν η Κομισιόν θέλει να σχολιάσει ε, και να αντιδράσει αυτά που ακούσαμε για τους νέους και το Ευρωπαϊκό Θελοντικό Πρόγραμμα. δεν ξέρω αν συζητήσατε στο Στρασβούργο όταν έγινε η εκδήλωση. Ε, η Λίντα θα παρουσιάσει τώρα μια άλλη ιδέα. Ευχαριστώ πολύ. Αναφέρεται στις τελευταίες ε, παρεμβάσεις για τη διακίνηση ανθρώπων και την εφαρμογή του νόμου. Η τελευταία έκθεση Europol έδειξε ότι στο επίκεντρο του προβλήματος ε, ε, είναι ένα δίκτυο που το αξιοποιεί το 90% των παράνομων μεταναστών. Ε, είναι σημαντικό λοιπόν να βρεθούν νόμιμοι διάβλοι. Μπορούν να γίνουν περισσότερα για την εφαρμογή του νόμου και για την προστασία των συνόρων έτσι. Ε, θα καταπολεμηθεί και το οργανωμένο έγκλημα. Η συνεργασία μεταξύ των οργανισμών της Ένωσης και τρίτων χωρών είναι σημαντική. Υπάρχουν πλατφόρμες συνεργασίας μεταξύ κρατών και οργανισμός Europol, Eurojust, αλλά είναι τεράστιο το πρόβλημα στις τρίτες χώρες και γι' αυτό χρειάζονται πιο πολλά πράγματα για αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών οργανισμών, τρίτων χωρών και κρατών μελών για την καταπολέμηση αποτελεσματικότερα του οργανωμένου εγκλήματος. Ε, τελευταία υπάρχει, έχει δημιουργηθεί το κέντρο ε, κατά της διακίνησης ε, ανθρώπων. Είναι σημαντικό να γίνει και αλλού και θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στη Μεσόγειο που εκεί υπάρχει μια πολυμερής ε, πλατφόρμα συνεργασίας πολλών χωρών. αυτό είχε αναφερθεί και στο Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας στα Βαλκάνια. Επίσης θα δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που θα δημιουργεί ένα αφήγημα ε, χωρίς να ε, θεωρεί ε, τους μετανάστες υπέτειους για κρούσματα βίας ε, υπάρχουν τέτοια αφηγήματα παντού. Ο στιγματισμός ως εγκληματιών των μεταναστών ε, έπαιξε πολύ κακό ρόλο. Θα πρέπει λοιπόν να είναι σαφές το αφήγημα. Δεν είναι οι, οι ε, παράνομοι οι μετανάστες, ε, δεν είναι οι εγκληματίες εκείνοι, αλλά ε, εκείνοι που τους εκμεταλλεύονται από το οργανωμένο έγκλημα. Ο η δεύτερη μου πρόταση είναι να δημιουργήσουμε μια βάση δεδομένων όπου θα υποβάλουν το βιογραφικό τους οι μετανάστες για να διαπιστωθεί αν έχουν δεξιότητες που χρειάζονται στις χώρες ε, που θέλουν να μεταναστεύσουν θα υποβάλλεται αίτηση στο κράτος μέλος, το κράτος μέλος θα ε, παληθεύει την ε, αίτηση, θα την επιβεβαιώνει και θα ενημερώνει αν υπάρχει ενδεχόμενο απασχόληση ε, από για το μετανάστη ανάλογα με γλώσσες, δεξιότητες κλπ. Είναι πιο σημαντικό να, βλέπω, ε, να, να ακολουθεί μια τέτοια διαδικασία και για το κράτος μέλος και για το μετανάστη. Θα πρέπει να ε, λαμβάνεται υπόψη και η βούληση του μετανάστη αλλά και οι ικανότητες ένταξης από τη χώρα μέλος. Έτσι θα είναι πολύ πιο διαφανής η διαδικασία εισόδου. Ο συνδικαλιστής ξέρω πόσο δύσκολο είναι να μπει κανείς στη σημερινή αγορά εργασίας. Ακόμα και οι μεδαποί δυσκολεύονται όταν πρόκειται για μετανάστες. Τα προβλήματα είναι ακόμα μεγαλύτερα αφού πρέπει να ξεπεράσουν γλωσσικούς φραγμούς, ε, δεν ξέρουν αν θα αναγνωριστούν οι δεξιότητες ε, και αυτό ε, δημιουργεί έλλειψη αυτοπεποίθησης. Οι χώρες υποδοχής θα πρέπει να δίνουν στους μετανάστες λοιπόν και καλή επιμόρφωση, ε, κατάρτιση για να μπουν στην αγορά εργασίας. Και έτσι περνώ σε ένα άλλο σημαντικό θέμα της ένταξης, ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας. Ε, θα πρέπει να αναγνωριστούν ε, τα προσόντα που έχουν ήδη. Πολλές φορές είναι υψηλή εξειδίκευση και δεν αξιοποιούνται γιατί δεν αναγνωρίζονται τα προσόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν ε, εκπαιδευτεί αλλού. Χρειάζεται ένα σύστημα ισοδυναμίας των διπλωμάτων, συστήματα πιστοποίησης που να αναγνωρίζονται από τη χώρα υποδοχής. Για να επιτύχει ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στον δημόσιο τομέα, στις δημόσιες υπηρεσίες δηλαδή. Ευχαριστώ. Ποιος θέλει να απαντήσει, να αντιδράσει σε αυτές τις τελευταίες δύο ιδέες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, λέει η κυρία Χιμένεθ. Μου φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η συνάντηση γιατί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ζητήματα όπως είναι το θέμα της μετανάστευσης, κάτι το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ τους απλούς ανθρώπους και τους νέους. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω για αυτήν την συνεδρίαση. Είναι πολύ καλό το ότι γίνεται και με την παρουσία και των δύο επιτροπών της ΑΦΕΤ και της ΔΕΒΕ. Αυτό το οποίο απαραίτητο εδώ πέρα να ενισχύσουμε είναι η αξιοπιστία της Ευρώπης. Αυτό είναι ένα ουσιαστικό θέμα γιατί εδώ παίζεται όλο το παιχνίδι γιατί οι πολίτες περιμένουν απαντήσεις και για την ασφάλεια και για την τρομοκρατία και την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών και της κρίσης των προσφύγων που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή στα μάτια των νέων διακυβεύει το κατά πόσο θα θεωρήσουν ότι αξίζει τον κόπο να αγωνιστούν για την Ευρώπη. Η Υπηρεσία Εξωτερικών, Εξωτερικής Δράσης έχει τονίσει την ε, ανάγκη αλληλεγγύης και προς τις χώρες που βρίσκονται έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μεταξύ των χωρών που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως είναι σημαντικό να ξέρουμε ποιο είναι το μήνυμα που θα δώσουμε στους νέους, κατά πόσο είμαστε σε θέση να συμφωνήσουμε μεταξύ μας σε ένα τόσο κέριο αλλά και δύσκολο θέμα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε <clears throat> το θέμα της ε, πηγής αυτών των ροών. Αυτό δεν μπορεί να επιληθεί από την Ευρώπη την ίδια. η Ευρώπη δεν μπορεί να τα λύσει όλα αυτά τα προβλήματα. Είναι προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν στις χώρες προέλευσης, στη ρίζα του προβλήματος. Και έχουμε το πρόβλημα των ε, διακινητών που χρησιμοποιούν τους ανθρώπους σαν να είναι εμπορεύματα και προσπορίζονται εκατομμύρια και εκατομμύρια. Πέραν των εκθέσεων που έχουμε κάνει και όλων αυτών που έχουμε τονίσει. Δεν έχουμε ασκήσει πραγματική πίεση για να αντιμετωπίσουμε <clears throat> το πραγματικό πρόβλημα που είναι ότι ασκείται αυτή τη στιγμή ένα παράνομο εμπόριο ανθρώπων. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να σταθούμε στο θέμα της διακίνησης ατόμων και επίσης να αντιμετωπίσουμε και τη ρίζα του προβλήματος, γιατί αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, μπορούμε να ζητάμε, να προσπαθούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, να ζητήσουμε το φεγγάρι και τα άστρα δεν θα πετύχουμε τίποτα. Χρειάζεται αλληλεγγύη και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορέσουμε να έχουμε μια κοινή θέση και να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Τελειώνει ο χρόνος. Δεν, είπα, δεν είδα κάποιον άλλο που θέλει να ε, πει κάτι. Ίσως κάποια τελικά σχόλια για, τα δύο αυτά, για τις δύο αυτές ιδέες. Η Λίντα πρώτα. <clears throat> Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να συζητήσουμε το αφήγημα το οποίο διαδίδει προς τους πολίτες η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί λένε ότι οι συμφωνίες που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μετανάστευση ότι είναι κάτι το οποίο γίνεται για το συμφέρον της. <clears throat> Αυτό όμως δημιουργεί μια αρνητική κατάσταση που οδηγεί τους νέους οι οποίοι περιμένουν μια απάντηση για από την Ευρωπαϊκή Ένωση να απογοητεύονται μπορεί η κατάσταση να βελτιωθεί στο μέλλον. Αλλά αν δίνεται σαν προτεραιότητα αυτές τις ε, συμφωνίες, αυτό σημαίνει ότι υποχωρεί σε σχέση με τις αξίες της Ευρωπαϊκή Ένωση και ασχολείται μονάχα με το θέμα της ασφάλειας. Αν δεν υπάρξει καλύτερη ασφάλεια και καλύτερη κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη στη γειτονιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν νομίζω ότι μπορούμε να βελτιώσουμε τη σχέση μας με τις χώρες της ε, νότιας όχθης της Μεσογείου και της Αφρικής. Όλα αυτά λοιπόν είναι η ουσία του προβλήματος. Είναι θέμα πολιτικής θέλησης για μένα. Και θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια συνεκτική στάση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ανδρέα. Θα ήθελα να απαντήσω στα προηγούμενα σχόλια Πράγματι, υπάρχει πρόβλημα με το ενότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να συνδυάσουμε τις προσπαθίες μας. Κατά κάποιο τρόπο είναι λογικό να υπάρχουν αποκλίνωσες ε, απόψη, όμως ε, το σύνθημά μα ε, είναι ενωμένη στην ποικιλομορφία. Πώς φτάνουμε λοιπόν σε αυτή την ενότητα. Νομίζω ότι μία από τι ε, λύσεις ε, και πάλι έγκυται στου νέους, γιατί ουσιαστικά συναντιούνται πιο εύκολα και δέχονται πιο εύκολα τις διαφορές μεταξύ των ανθρώπων. Λοιπόν, πρέπει να συνεχίσετε να επενδύετε σε προγράμματα για την νεολαία, γιατί όταν εμπλέκετε τους νέους, τους δίνετε και νόημα. Παραδείγματο χάρη, η σημερινή εμπειρία είναι πολύ σημαντική για μα, προκειμένου να δούμε ότι μα ακούνε και μάλιστα είμαστε ακόμη και πιο ενθουσιώδει όταν βλέπουμε ότι θα γίνουν πραγματικότητα κάποιες από αυτέ τι ιδέε. Ας μην ξεχνάμε ότι ένα οίκος χωρίς ενότητα είναι οίκος χωρίς δύναμη, χωρίς εξουσία. Έτσι λοιπόν ας δώσουμε δύναμη σε αυτόν τον οίκο. Ο Ματέους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που συμφωνείτε. Χαιρόμαστε που ακούμε ότι σας αρέσουν οι ιδέες μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι ακόμη πιο ισχυρή και να δείξει ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να συνεργαστούν προκειμένου να επιλύσουν το μεταναστευτικό πρόβλημα. Καθώς εμείς οι τρεις εκπροσωπούμε τη μεγαλύτερη εκδήλωση της νεολαίας και εκπροσωπούμε την νεολαία της Ευρώπης, νομίζω ότι σας δείξαμε ότι θέλουμε μια Ευρώπη που να στέκεται ενωμένη, να είναι ελεγγύα και θέλουμε οι νέοι να έχουν φωνή και φυσικά να ακούγεται η φωνή τους. Σας ευχαριστώ. Να δούμε αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να αντιδράσει. Το πολύ δύο λεπτά παρακαλώ. Μαρία Δεπαόλης, παρακαλώ. Δεν ξέρω που κάθεστε. Εκεί κάτω. Ευχαριστώ Μαρία. Ε, μετά Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήδη η ΔΕΦΚΟ αντιμετωπίζει τις ε, αιτίες της μετανάστευσης. Μπορώ να αναφέρω κάποια παραδείγματα εφαρμόζουμε δράσεις για να δώσουμε ε, εξουσίες, αρμοδιότητες στην νεολαία σε κάποιες χώρες, σε χώρες για να μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Εφαρμόζουμε προγράμματα στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και αναλύουμε τις δυνατότητες να βελτιώσουμε την αγορά εργασίας και να αποφύγουμε τις αναντιστοιχίες μεταξύ της ε, εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας. Επίσης, ε, θα έχουμε να αναγνωρίζονται τα προσόντα στις χώρες εταίρους, προκειμένου να ενθαρρύνουμε την κινητικότητα μεταξύ των χωρών. Και φυσικά σε ό,τι αφορά τις αιτίε, ε, δεν ε, πρέπει να εστιαστούμε μόνο αυτό. Πρέπει ουσιαστικά να δούμε ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι από την παιδική τους ηλικία. Τα σημερινά παιδιά θα γίνουν η επόμενη γενιά μεταναστών. Και βλέπουμε πολλά παιδιά μετανάστες να έρχονται στην Ευρώπη ασυνόδευτα. Και είναι σε πάρα πολύ ευάλωτη κατάσταση. Επομένως, έχουμε μία σειρά δράσεων στην Κομισιόν που στοχεύουν στο να διασφαλίσουν τη συνεκτικότητα, αλλά κάνουμε και μία αποτίμηση άλλων πολιτικών που έχουμε εφαρμόσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης συνεργαζόμαστε με το ΕΚΟ, το Γραφείο Ανθρωπιστικής Βοήθειας, για να προσφέρουμε εκπαίδευση, υπηρεσίες υγείας και όλες τις βασικές υπηρεσίες που είναι απαραίτητες στους πρόσφυγες. Αυτά είναι μόνο κάποια παραδείγματα. Αν χρειάζεται περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να απευθυνθείτε απευθεία σε εμά. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω και τους προσκεκλημένους μας σήμερα. Βλέπετε ότι τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπαθούν να βρουν λύσεις για το μεταναστευτικό, αλλά πολλές φορές μπλοκάρουν τα κράτη-μέλη. Ε, υπάρχουν πολλά δύσκολα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, η κοινή γνώμη και ε, εδώ βέβαια καλό είναι που μας ενημερώσατε, αλλά καλό είναι να διαμορφώνεται και συνένεση μέσα από τη δική σας προσπάθεια και στις χώρες μέλη. Ε, θα πρέπει να δοθεί μάχη σε κάθε επίπεδο για μια πιο συνεκτική ευρωπαϊκή πολιτική. Να ευχαριστήσω με πάρα πολύ λοιπόν τους προσκεκλημένους μας που ήρθαν με τις ιδέες τους εδώ σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι καλή ιδέα ότι ακούσαμε περισσότεροι ε, από διάφορες επιτροπές τις προτάσεις σας. Ελπίζω ότι ε, στην επόμενη συζήτηση θα ε, ληφθούν υπόψη και άλλες ιδέες για τη μετανάστευση. Προχωράμε τώρα στο σημείο 13 κοινή